διαταξή είναι η προφορική ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα στι εμπορικέ διαπραγματεύσει Ευρωπαϊκή Ένωση και Βιετνάμ. Από την Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου και θα δώσω το λόγο στον συντάκτη τη ερώτηση, τον κύριο Λάγκα, για πέντε λεπτά. Σα ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, κυρία Επιτροπέ. Τι επόμενε εβδομάδε ε, στις του ο Πρωθυπουργό του Βιετνάμ θα μεταβεί στις Βρυξέλλες ε, προκειμένου να υπογράψει την εμπορική αυτή ε, συμφωνία η οποία και θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή συμφωνία η οποία έχει ε, αποτελέσει το αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιετνάμ με σαφή και ασύμετρη πρόγραμμα μείωση των δασμολογικών επιβαρύνσεων. Συμφωνήσαμε για νέα πρότυπα, 169 GIs έχουν γίνει δεκτά από το Βιετνάμ για τα θέματα δημοσίων προμηθειών δεν υπάρχει συμφωνία, αλλά σε γενικές γραμμές υπάρξει, υπάρχει, ε, πραγματικά, υπάρχουν πλέον ίσοι όροι επί των οποίων συμφωνήσαμε. Θα είναι λοιπόν αξιοσημείωτη αυτή η εμπορική συμφωνία και στο προήμιο γίνεται σαφώς αναφορά στην Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ του 42 και του 48. Στην εμπορική λοιπόν συμφωνία γίνεται σαφής αναφορά στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην εξασφάλιση το, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτών. Και άρα αυτή η εμπορική συμφωνία και η συνεργασία ε, συνεργασίας η οποία επιτεύχθη το 2012 αποτελεί λοιπόν έτσι ένα νόμιμο σύνδεσμο ένα νομικά δεσμευτικό σύνδεσμο. Και έτσι λοιπόν αυτή η Συμφωνία Εταιρική Σχέση και Συνεργασία αποτελεί κάτι που έχει σημασία και για την εμπορική συμφωνία. Και γι' αυτό λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι πιστεύω συμφωνούμε όλοι ότι πρώτα θα είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και μετά ε, θα πρέπει να συνδέσουμε άρρηκτα το εμπόριο με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μπορώ να φανταστώ οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία που δεν γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και επίσης ε, στην συμφωνία τι που προσπογράφει και το Βιετνάμ ε, γίνεται ακριβώς τέτοια σύνδεση μεταξύ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της, ε, του ανοίγματο της αγοράς. Ένας αυτοματισμός. Άρα τα ανθρώπινα δικαιώματα συγκαταλέγονται στα βασικά θέματα του εμπορίου. Και κοιτώντα λοιπόν το Βιετνάμ, διαπιστώνουμε όλοι ότι είναι μια πολύ δυναμική χώρα σε φάση μεταμόρφωση και αντιμετώπιση προκλήσεων ασφαλώς σε αυτή τη φάση της μεταρρύθμισης. Και πολλά θέματα ανθρωπινών δικαιωμάτων θα πρέπει να επισημανθούν, ιδιαίτερα στο θέμα τη ελευθερία έκφραση. Και ω μέσο, ασφαλώ, ω μέσον, στα πλαίσια των διαφόρων ρητρών ε, στην εμπορική συμφωνία συνδέεται και ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και εδώ είναι λίγο το πρόβλημα. Το θέμα του πώς το θέμα του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί να βελτιωθεί προκειμένου στην πράξη να έχει μεγαλύτερη ε, επιρροή. Και εδώ θα ήθελα σε πέντε ζητήματα να τονίσω το κατά πόσο χρειάζεται βελτίωση. Καταρχάς, ε, του ορισμού των, ε, του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Χρειάζονται συγκεκριμένα milestones, ε, στόχοι δηλαδή. Κατά δεύτερον, πώς μπορούμε να πετύχουμε να εμπλέξουμε καλύτερα την κοινωνία των πολιτών στο διάλογο αυτό. Για να συμμετάσχει και η κοινωνία των πολιτών υπάρχει το Civil Society Forum και άλλες οργανώσεις και τα ανεξάρτητα συνδικάτα ενδεχομένω να αναπτυχθούν από τον διάλογο αυτό. Μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα υπάρχουν σαφείς κανόνες και ηλική υποστήριξη προκειμένου σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μέσα από την κοινωνία των πολιτών. Κατά τρίτον, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τις υπηρεσίες εξωτερικής δράση, αλλά και σε ό,τι αφορά συγκεκριμένε συγκεκριμένες προκειμένου να υπάρχει πραγματικά συνοχή από πλευρά της Ένωσης. Κατά τέταρτον, τι γίνεται με την αξιολόγηση του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μπορούμε να βάλουμε πιο σαφείς δείκτες και πέμπτον, η διαφάνεια, αγαπημένο μας θέμα. Και στον ε, διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να ενισχύσουμε την πτυχή της διαφάνειας. Αυτά είναι λοιπόν κάποια ερωτήματα για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τον διάλογο για ανθρώπινα δικαιώματα σε ό,τι αφορά και το Βιετνάμ, αλλά και σε ό,τι αφορά και την εμπορική στρατηγική και τις μελλοντικέ ε, συμφωνίες. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ, λέει και η Πρόεδρος, λέει η Πρόεδρος από τον κύριο Λάγκα. Και τώρα η κυρία Μάλμστρομ, εξ ονόματος της Επιτροπής. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι η Κομισιόν έχει αναλάβει να προάγει ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις συμφωνίες ε, με τρίτες χώρες και γι' αυτό το λόγο έχουμε οργανώσει τον ε, Μάιο μια συζήτηση των άμεσα ενδιαφερομένων και το έγγραφο που δημοσιεύτηκε επισημαίνει ότι πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί η κατάσταση ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εκεί υπογραμμίζεται και η δική μας συνδέσμευση για την συμπερίληψη και της κοινωνίας των πολιτών. Θέλω λοιπόν να επισημάνω ότι θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν ενταχθεί σε αυτή τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Βιετνάμ και με στόχο να συμπεριληφθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην τελική μορφή της ε, συμφωνίας. Περαιτέρω στόχος είναι να μην υπάρξουν αρνητικές συνέπειες και αυτό το έχω συζητήσει με τους αρμόδιους υπουργούς. Ε, στο προήμιο αναφέρεται ότι το Βιετνάμ δεσμεύεται να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης υπάρχει ε, και μία νομική σχέση ανάμεσα στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ε, ε, φαρμογή των εμπορικών συμφιών. Αναφέρεται ότι οι συμφωνίε που ισχύουν είναι και η FTA και μπορούμε να λάβουμε μέτρα οποτεδήποτε θεωρούμε ότι υπάρχει παραβίαση της συμφωνίας. Εξάλλου η συμφωνία FTA ελεύθερο εμπορίου δηλαδή, ε, περιλαμβάνει και πολλές άλλες νομικές λεπτομέρειες, γιατί με τον τρόπο αυτό ενισχύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου ε, στο Βιετνάμ. Όσον αφορά τα εργατικά δικαιώματα, αυτό είναι ένα ε, πολύ φιλόδοξο κεφάλαιο Βεβαίως ε, θα πρέπει να επικυρωθούν οι συμφωνίες ε, που, που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο του ILO να υπάρχουν ε, προγράμματα αδιάβλητα και δίκαια. Στο Βιετνάμ θα συνεχίσουμε να έχουμε παρακολούθηση των εφαρμοζομένων, διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μετά από κάποιες εβδομάδες θα ξαναγίνει μία συνάντηση και έχουμε και επίση το Ευρωπαϊκό Εργαλείο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, όπω όλοι πολύ καλά γνωρίζετε. Οι δεσμεύσει μα θα παρακολουθούνται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Βιετνάμ μέσα από ένα θεσμό. Συστάθηκε, συστήθηκε ακριβώ για αυτό το σκοπό και μέσα από αξιολογήσει εκ των υστέρων. Εγώ λοιπόν είμαι ακράδαντα πεπισμένη και νομίζω ο κ. Λάγκε το είπε και αυτό το ίδιο, ότι η απελευθέρωση του εμπορίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν και πρέπει να συμβαδίζουν. Είναι ανακοίνωση για το εμπόριο και τι επενδύσει που δημοσίευσε πριν από κάποιε εβδομάδε η Κομισιόν καθιστούν σαφέ ε, ότι αυτά θα πρέπει να ισχύουν για όλου, του καταναλωτέ, ε, του ελεύθερου επαγγελματίε, τι μικρομεσαίες επιχειρήσει και προφανώ και του πιο φτωχού στι αναπτυσσόμενες χώρε. με στόχο την ε, ευημερία, την ανάπτυξη, όλα όμω με υπευθυνότητα. Άρα δηλαδή η εμπορική μα πολιτική πρέπει να περασπίζεται τι δικέ μα μας αξίες, να είναι αποτελεσματική, πρέπει να είναι διαφανής, ανοιχτή στο δημόσιο έλεγχο. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολύ σημαντικά στο πλαίσιο αυτή τη εμπορική στρατηγική. Η Κομισιόν επιθυμεί να διασφαλίσει ότι η εμπορική πολιτική συμβάλλει ε, στην ε, στήριξη, στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στι δύο πλευρέ, σε συνδυασμό και με άλλε πολιτικέ, στην εξωτερική πολιτική, πολιτική ανάπτυξης, ανάπτυξης και ούτω Η ισορροπία ανάμεσα στην αφοσίωση και τι προποθέσει engagement και conditionality, ξέρετε ότι η Κομισιόν θεωρεί η πρώτη πολιτική είναι πολύ καλύτερη από τον εφαρμόζονται μόνο προϋποθέσεις. Η αφοσίωση, η δέσμευση μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε ε, διόδους ε, διαλόγου με όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους και έχουμε στόχο να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα κανάλια για να επιτύχουμε αλλαγή επιτόπου στο Βιετνάμ. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεισφορά σας και να είστε σίγουροι ότι ε, μόλις ολοκληρωθεί η συμφωνία θα σας ενημερώσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και εμείς ε, και τώρα για δύο λεπτά ο κύριος Φίσας. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, μετά από την ε, υπογραφή συμφωνίας το 2012 μεταξύ Βιετνάμ και Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάσαμε σε μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με μια κομμουνιστική χώρα. Έχει μεγάλη σημασία αυτή η εμπορική συμφωνία. Πιστεύουμε ότι το ΑΕΠ ε, αυτής της χώρας θα αυξηθεί κατά 6% και θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις εμπεδίσεις. Πρόκειται για ένα δεσμευτικό πλαίσιο που περιλαμβάνει ρήτρε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έτσι ώστε να ε, διέπονται σωστά αυτές οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιετνάμ. Μετά από 25 χρόνια αποκατάστασης των ε, διπλωματικών σχέσεων ασχολούμαστε ακόμα με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ. Υπάρχει η θανατική ποινή που υπάρχει ακόμα, υφίσταται ακόμα ε, δίωξη ακτιβιστών και έλλειψη ανεξιθρησκείας. Θα πρέπει λοιπόν να εξαλειφθούν αυτές οι πρακτικές. Μην ξεχνάμε όμως ότι το Βιετνάμ κάνει βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, είναι μέλος του ΟΗΕ που το 2014 ψήφισε κατά των βασανιστήριων παγκοσμίω. Είμαι ο καλύτερος φίλος μας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στα πλαίσια της ΑΣΕΑΝ και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ευχαριστούμε για ένα μισή λεπτό κυρία Μόσκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Η εμπορική συμφωνία που θα ολοκληρωθεί στις 2 Δεκεμβρίου μεταξύ Βιετνάμ και Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μεγάλη σημασία. Όχι μόνο για τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΣΕΑΝ και την εμπορική μας πολιτική. Είναι μια στρατηγική συμφωνία, γι' αυτό το λόγο, αλλά όπως είπε και ο πρόεδρος Λάγκε, και για την ποιότητα των διαπραγματεύσεων. Γι' αυτό είναι ένα πρότυπο για μελλοντικές συμφωνίες και γι' αυτό θα πρέπει να εποπτεύσουμε πολύ προσεκτικά όλες τις επιπτώσεις, ιδιαίτερα για την ανάπτυξη της, για το, στο κεφάλαιο της βιώσιμης ανάπτυξης, που έχει σημασία και για την εμπορική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι' αυτό υποβάλαμε αυτό το ερώτημα στην Επιτροπή για να έχουμε περισσότερες πληροφορίες και πιο συγκεκριμένες. Και ευχαριστούμε την Επίτροπο γιατί σήμερα ε, μοιράστηκε μαζί μας σημαντικά στοιχεία. Πιστεύουμε ότι υπάρχει μια βελτίωση της εποπτείας σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τις χώρες ε, με τις οποίες συνάπτουμε συμφωνίες και για να υπάρχουν νέα πρότυπα αξιολόγησης και επιπτώσεων με τη συμμετοχή και της κοινωνίας των πολιτών στις διαπραγματεύσεις. Θεωρούμε ότι οι εμπορικές ε, συμφωνίες θα πρέπει να αποτελέσουν ένα μέσο βελτίωσης και των κοινωνικών συνθήκων διαβίωσης. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να συνάπτονται συμφωνίες αν δεν λαμβάνουν υπόψη αυτή τη διάσταση του ζητήματος. Ε, στραπάτη για ένα λεπτό. Πρόκειται για μια δυναμική χώρα, νέα χώρα, και κυρίως για μια χώρα που δεν ναι, περιμένει να έρθουν οι θέσεις εργασίας, αλλά δημιουργεί θέσεις εργασίας. Αυτό το διαπιστώνουμε επανελειμμένα. Υπάρχει κομμουνιστική κυβέρνηση, κομμουνιστική και κομμουνιστικό κόμμα, αλλά δεν ε, είναι... Δεν ακολουθεί τις συνθήσεις οδούς των σοσιαλιστών ο κόσμος μπορεί να εκφραστεί όπως θέλει όσο δεν ενοχλεί τα, τις αρχές. Και εδώ μπαίνει στο παιχνιδί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και πιστεύω ότι είναι λάθος να είμαστε πάντα να προδιαγράφουμε τι θα πρέπει να συμβεί σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει να κοιτάμε και να αναλύουμε τι συμβαίνει. Σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο χρειαζόμαστε ανθρώπους που μπορούν να σκεφτούν και μπορεί κανείς να σκεφτεί και να διαπραγματευτεί μόνο αν υπάρχουν ε, ανθρώπινα δικαιώματα για λόγους ανάλυσης για τα δικά τους ε, συμφέροντα θα πρέπει να τους εξηγήσουμε ότι θα πρέπει να προσεγγίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ η κυρία Σχάκε για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Οι φιλελεύθεροι καλωσορίζουν το γεγονός ότι αυτή η πρώτη τέτοιου είδους ε, συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιετνάμ με μια αναπτυσσόμενη χώρα έχουν ολοκληρωθεί και πιστεύουμε ότι είναι καλή συμφωνία. Το εμπόριο ως γενικότερο πλαίσιο της γενικότερη ατζέντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα συγκεκριμένο εργαλείο όπου παίζει ηγετικό ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τις πολιτικές ανάπτυξης. Βλέπουμε ότι οι πολίτες όλο και πιο πολλοί συμμετέχουν στη συζήτηση αυτή. Είναι ευπρόσδεκτο αυτό και ο κόσμος στην Ευρώπη είναι σαφής. Θέλουν στην κορυφή των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ε, πολιτικής της εξωτερικής της Ένωσης να είναι τα τρόπινα δικαιώματα. Πιστεύω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και ευκαιρία και ευθύνη να προωθήσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελεί μόχλευση. Γιατί ακούγοντας τη δημόσια συζήτηση που διεξαγάγεται, ε, πιστεύω ότι σε κάποιες περιπτώσεις είναι κάπως υπέρμετρες οι φιλοδοξίες του κόσμου σε ό,τι αφορά τον ρόλο του εμπορίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει όμως αυτά να αποτυπώνονται στην ε, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πέρα από την αναμενόμενη, το αναμενόμενο έναυσμα στην ε, ανάπτυξη και στην οικονομία του Βιετνάμ, θα ήθελα να ξέρω ποια είναι τα βραχιοπρόθεσμα μέτρα τα οποία αναμένονται. Πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο θέμα του εμπορίου και πώς θα υπάρξει παρακολούθηση μετά τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας. Πολλά θα πρέπει να βελτιωθούν στο Βιετνάμ η ελευθερία έκφρασης του συναθρίζεσθε. Όλα αυτά είναι υπό έλεγχο, υπό πίεση. Δυστυχώς εξυλοδαρμοί και ε, βασανιστήρια τακτικά λαμβάνουν χώρα και οι μειονότητες πλήττονται ιδιαιτέρως. Κλείνοντας λοιπόν και πάλι, πρέπει να επαναλάβω ότι όλες αυτές οι προκλήσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω του εμπορίου. Θα πρέπει να αναπτύξουμε τον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα πρέπει να δούμε λοιπόν ποια θα είναι, ποιος θα είναι ο αντίκτυπος της εμπορικής αυτής συμφωνίας στα ανθρώπινα δικαιώματα στο Βιετνάμ. Ευχαριστώ για 1,5 λεπτό. Η κυρία Σάντσος έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Επιτροπή έφτασε σε μία συμφωνία με το Βιετνάμ. Αυτό δεν μας ε, εκπλήσει, αλλά δεν ελήφθησαν υπόψη οι συστάσεις ε, του Κοινοβουλίου και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Δεν λάβαμε υπόψη τις συστάσεις του ΟΗΕ περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βεβαίως ε, ε, περιλαμβάνουμε κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά ξέρουμε άρα ωραία λόγια και τίποτα άλλο. Τι εγγύσεις υπάρχουν ότι τα μέρη θα ε, ανταποκριθούν προς τις υποχρεώσεις τους. Θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με την ισότητα των δύο φύλων. Η Εμπορική Επιτροπή, η Εμπορική Συμφωνία δεν περιλαμβάνει διατάξεις για την ισότητα των δύο φύλων και ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την πλήρη ατιμορρησία των μεγάλων κοινοπραξιών. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό θα ήταν αποτυχία της ευρωπαϊκής ε, πολιτικής με δραματικές συνέπειες ιδιαίτερα για, τα, για τους ανθρώπους. Η κυρία Κέλλερ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ το να προστατεύει κανείς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή είναι η ουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Και θα έπρεπε να είναι και το επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Εμπορικής Πολιτικής. Ε, στο Βιετνάμ ε, δεν γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε υπάρχει και ελευθερία τύπου, απαγορεύονται τα πολιτικά κόμματα, τα συνδικάτα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη νέα της εμπορική στρατηγική, η οποία φέρνει μπροστά στο προσκήνιο τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το θέμα είναι όμως πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά στην εμπορική πολιτική. Και εκεί λοιπόν ε, κάτι πρέπει να γίνει στο Βιετνάμ. Δεν έχουν γίνει ακόμα εκτιμήσεις ε, για τις επιπτώσεις των εμπορικών συμφωνιών. Έχουμε αρκετά ερωτηματικά, κυρίως όσον αφορά την, ε, και την προστασία των επενδυτών. Σε αυτές τις ε, συμφωνίες δεν βλέπουμε να υπάρχει το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι λοιπόν σημαντικό να δούμε πολύ συγκεκριμένα τι μπορούμε να πετύχουμε με το εμπόριο στο Βιετνάμ, κυρίως τα ανθρώπινα δικαιώματα. Καλά τα λόγια, αλλά μετά από τα λόγια πρέπει να ακολουθήσουν και τα έργα. Ευχαριστώ πολύ για ένα λεπτό Ευχαριστώ, κυρία Μπεγκίν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ είναι τραγική. Ε, υπάρχει ένα μόνο κόμμα το οποίο καταπιέζει όλε τι ελευθερίε, την ελευθερία του συνέρχεστε, τη έκφραση, Όλα λοιπόν παραβιάζονται συστηματικά. Υπάρχουν βασανιστήρια και επίση και εξαναγκαστική εργασία για αγαθά προς εξαγωγή. Και τι κάνει η Ευρώπη, αποφασίζει να τους επιβραβεύσει με μία μια συμφωνία ελεύθερων ανταλλαγών που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ε, μέσο ε, άσκησης πίεσης για να επιτύχουμε πραγματικές αλλαγές. Για άλλη μια φορά λοιπόν ε, συνάπτουμε συμφωνίες με δικτάτορες και χρησιμοποιούμε προς αυτού την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Οι δικοί μας οι Γεωργοί θα έχουν 80 εκατομμύρια ρύζι από το Βιετνάμ που θα έρθει στις δικές μας αγορές από την Καμπότζη, από την Μιανμάρ. Αυτή λοιπόν είναι η εμπορική ευρωπαϊκή πολιτική που βασίζεται σε αξίες. Εσείς έτσι πιστεύετε, εγώ δεν το πιστεύω αυτό, κυρία Επίτροπε. Σας ευχαριστώ. Ένα μισή λεπτό, κύριο Φιέλνερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την ε, Επίτροπο. Ολοκληρώθηκε λοιπόν αυτή η διαπραγμάτευση μετά από τρία χρόνια μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Βιετνάμ. Είναι σημαντική λοιπόν αυτή η συμφωνία για το Βιετνάμ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η Ευρωπαϊκή Ένωση, η πιο σημαντική μετά την Κίνα. Και ελπίζουμε λοιπόν να επιτρέψει αυτή την ανάπτυξη τη χώρα. Είμαι πεπισμένη ότι είναι ο καλύτερο τρόπο αυτή η συμφωνία για να εξέλθει από τη φτώχεια η χώρα. Και αυτό το βλέπουμε και στην Σουηδία. Υπάρχει η δυνατότητα να δοθούν λοιπόν τέτοιες ευκαιρίες και σε άλλες αγορές σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιοι που διατείνονται ότι δεν υπάρχει αυτοματισμός και ότι το εμπόριο είναι απειλή για τα δικαιώματα. Αυτό δεν στέκει, γιατί διαπιστώνουμε τι συμβαίνει. Οι Βιετναμέζοι επιθυμούν αυτή τη συμφωνία και πρέπει να δούμε λοιπόν τι θα συμβεί δεν μπορούμε λοιπόν να διατηνόμαστε ότι δεν θέλουν αυτή τη συμφωνία. Τη στιγμή που την θέλουν είναι πολύ σαφέ οι θέσει. σαφείς λοιπόν οι θέσεις του και σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και σε ό,τι αφορά το περιβάλλον. Και εδώ πέρα θεωρώ ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε και τις δικαιολογίε που χρησιμοποιούνται. Πάντα υπάρχουν δικαιολογίε για να υπάρχουν εμπόδια στις ανταλλαγές αυτές και στις συναλλαγές αυτές. Και είδαμε λοιπόν τι είπαμε και από τη Βερμανία η Πρωθυπουργό σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα, σε ό,τι αφορά το Πακιστάν, σε ό,τι αφορά τη Μαλάλα. Ήταν κατά. Τώρα είμαστε λοιπόν κατά του Βιετνάμ, γιατί εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι είναι καλύτερα, ότι ξέρουμε καλύτερα τι είναι καλό για τις χώρες αυτές και όχι αυτές οι ίδιες. Αυτό είναι μια καινούργια τάση. Ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Μάρτιν για 1,5 λεπτών. Ευχαριστώ Πρόεδρα και καταρχάς να πω ότι συμφωνώ με τον κύριο Λάγκα ότι είναι πάρα πολύ καλή αυτή η συμφωνία για οικονομικούς όρους και για την Ένωση και για το Βιετνάμ και θα σημαίνει ανάπτυξη και για τις δύο περιφέρειες. Κατά πόσο είναι τέλεια τώρα η κατάσταση στο Βιετνάμ. Όχι. Απέχει παρασάγκας, όπως είπαν και πολλοί συνάδελφοι. Κατά πόσο όμως θα βελτιωθεί η κατάσταση με τη συμφωνία αυτή. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Και εδώ συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η συμμετοχή, η δέσμευση στη διαδικασία αυτή θα βελτιώσει την κατάσταση αυτή. Χάρη στη συμφωνία λοιπόν αυτή θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τους Βετναμέζους και ελπίζουμε να υπάρξει μια συμβουλευτική ομάδα στο εσωτερικό της χώρας για να συμμετάσχει και η κοινωνία των πολιτών. Να υπάρχουν τακτικές ε, αναφορές για την κατάσταση και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κατάσταση για τα εργασιακά δικαιώματα να βεβαιωθούμε ότι τα σχετικά, οι σχετικές προδιαγραφές εφαρμόζονται και τηρούνται, ότι θα υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Αλλά όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν χωρίς τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου, χωρίς την ε, Συμφωνία Συνεργασίας. Δεν έχουμε βάση λοιπόν συνεργασίας χωρίς αυτές τις συμφωνίες. Είναι καλό λοιπόν και για την ανάπτυξη αλλά και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, η κυρία Κέρλινγκ. Σα Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα εξελίσσεται, δεν προκύπτει. Δεν προκύπτει επειδή απλά μια συμφωνία έχει επικυρώσει τις ε, διεθνείς ε, συμφωνίες ε, ή επειδή βομβαρδίζεται από αιτήματα από δυνάμει εταίρους. Ε, και αυτά εξελίσσονται όπως σας είπα. ΑΣΕΑΝ είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Βιετνάμ αποκτά μεγαλύτερη σημασία στην ΑΣΕΑΝ λόγω της οικονομίας του. Έτσι λοιπόν χαιρετίζω αυτή τη συμφωνία και πιστεύω ότι η συμφωνία αυτή θα βγάλει τους ανθρώπους από τη φτώχεια στο Βιετνάμ και θα τους δώσει τη δυνατότητα ε, να να προωθήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα τους. Εγώ ε, παρακολουθώ το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ και μερικές φορές εκνευρίζομαι και απογοητεύομαι. Χαίρομαι όμως που επιτέλους αυτή η συμφωνία θα ολοκληρωθεί. Ας είμαστε επικοδομητικοί, να συνεχίσουμε το διάλογο, να προσφέρουμε ε, στήριξη στην κυβέρνηση μέχρι η ε, συμφωνία αυτή να γίνει επιτυχημένη. Κυρία Γκέρλινγκ, δέχεστε μπλε κάρτα από τον κύριο Φωνσίνη. Τη δέχεστε. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ ε, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω τη συνάδελφό μας την κυρία Γκέρλινγκ ε, το εξή. Ε, το θέμα των αυστηρών προϋποθέσεων. Αυτό θα πρέπει να το συμπεριλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη στρατηγική της με τις αναπτυσσόμενες χώρες, με όλες συμπεριλαμβανομένου και του Βιετνάμου. Έχετε 30 λεπτά για να πατήσετε κυρία Γκέρλινγκ. Δεν κατάλαβα. Λυπάμαι, αλλά δεν κατάλαβα. Τι είπατε, στα αγγλικά ρώτησε ο μιλητής, στα αγγλικά παντά η κυρία, ξέρετε, θέλετε να μιλήσετε πάλι, να ξαναρωτήσετε. Ξανά. Η ερώτηση είναι η εξής. Μία πολιτική αφοσίωσης, δέσμευσης και προϋποθέσεων. Μια τέτοια πολιτική θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις σχέσεις που αναπτύσσει με τις αναπτυσσόμενες χώρες ε, και με το Βιετναμ. Λυπάμαι πολύ, αυτά τα αγγλικά δεν τα καταλαβαίνω, λέει η ε, Ευρωβουλευτής, επίσης τα αγγλικά, απορρίπτει την ερώτηση. Για δύο λεπτά δίνω το λόγο στην κυρία Λόχπιλε. Κυρία Επίτροπε, Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου στο Ανόη αυτό το μήνα είδα μία πρωτεύουσα με όλο και πιο ζωντανή οικονομία ε, που προσπαθεί να επιτύχει τους στόχους της χιλίτιας. Άκουσα όμως και για την ε, έλλειψη συνδικάτων, μεγαλύτερη καταπίεση. Η χώρα είναι 175η από τις 180 στον κατάλογο και στον δίκτυο για την ελευθεροτυπία. Ε, οι αλλαγές δεν προκύπτουν αυτόματα και δεν οδηγούν αυτόματα σε μια κοινωνία ε, με ανισότητες, σε μια κοινωνία με παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε μια κοινωνία με ισχυρά ε, εργατικά δικαιώματα. Γι' αυτό λοιπόν χαιρετίζω το ότι η Επιτροπή ήδη το 2012 δεσμεύτηκε ε, να προβαίνει ε, σε αξιολόγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάτι που εκφράζεται στο πρόγραμμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας. Τον Απρίλιο του 2014 το Κοινοβούλιο κάλεσε την Κομισιόν το συντομότερο δυνατόν να προβεί σε αξιολόγηση της κατάστασης των ανθρωπίων δικαιωμάτων. Ε, παρά λοιπόν τις επιστολές και την οξύτατη κριτική που ασκήθηκε από τον διαμεσολαβητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και η Κομισιόν αρνήθηκε να δεχτεί αυτή τη σύσταση. Λόγος, ε, δικαιολογία που ε, αναπτύχθηκε ήταν η έλλειψη χρόνου. Η Κομισιόν όμως ε, δεσμεύτηκε να συμπεριλάβει μία αξιολόγηση της κατάστασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην επόμενη προβλεπόμενη αξιολόγηση. Ήδη εφέτος το καλοκαίρι έχουν επισημηθεί οι αντικές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα και ε, πολλοί ζητούν και εξάντε και εξπόστα την αξιολόγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εγώ δεν πιστεύω ότι οποιαδήποτε δικαιολογία θα είναι επαρκής. Η Κομισιόν αυτό που πρέπει να κάνει είναι να προβεί σε μια ουσιαστική εμβρητή αξιολόγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο κύριος Κοράου, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, να χαιρετήσω και την Επίτροπο άκουσα τη συζήτηση και δεν ε, συμφωνώ με αυτή τη γενική ευτυχία που επικρατεί ως προς τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών ε, με το Βιετνάμ. Αυτή η αγάπη για το νέο φιλελευθερισμό σημαίνει ότι εθελοτυφλούμε ως προς τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι ε, πολύ σοβαρές. Βρίσκεται το Βιετνάμ στην 175η θέση ως προς την ελευθερή, ελευθεροτυπία. Ο, και η κυβέρνηση χρησιμοποιεί χούλιγκαν για να καταστήλουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει λοιπόν ε, να προβούμε στη βελτίωση, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε μέσω μιας εμπορικής συμφωνίας, ούτε με μια εταιρική σχέση γιατί βλέπουμε ότι ε, δυστυχώς επιδεινούνται η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. πρέπει να γυρίσουμε σελίδα όταν μιλάμε για αυτές τις συμφωνίες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριάς έχει μπλε κάρτα νομίζω. Έχει το λόγο, με συγχωρείτε. Το εξή σοβαρό ζήτημα στην Ολομέλεια. Το έχω θέσει και δεύτερη φορά. Η Ολομέλεια είναι για να μπορούμε να συμμετέχουμε στις συζητήσεις αφιερώνεται αυτή η εβδομάδα του στρασβούργου στην ολομέλεια. δεν μπορούμε να έχουμε ταυτόχρονα συνεδριάσεις των επιτροπών και ιδίως συνεδριάσεις και ψηφοφορίες σε επιτροπές. αυτή τη στιγμή 7 η ώρα καλούμε να συμμετάσχω σε ψηφοφορία σε κοινή συνεδρίαση της ΛΥΜΠΕ και της πέτη για ένα σοβαρό θέμα που είναι το frontex. διαμαρτύρομαι διότι εγώ θέλω να συμμετάσχω και στη συζήτηση δεν μπορεί λοιπόν το πρόγραμμα των επιτροπών να μας αφαιρεί το δικαίωμα συμμετοχής στην ολομέλεια. παρακαλώ να μεταφέρετε αυτό το θέμα στον κύριο πρόεδρο στον κύριο Σούλτς και να επισημανθεί στους προέδρους των επιτροπών ότι αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα ολομέλειας και όχι ψηφοφοριών σε επιτροπές. οι ψηφοφορίες στις επιτροπές άλλη εβδομάδα στις βρυξέλλες. ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και σημειώνουμε λοιπόν τα σχόλιά σας και θα τα διαβιβάσουμε στον κύριο Σούλτς και θα συνεχίσουμε λοιπόν τώρα τη συζήτηση. Για ένα μισό λεπτό τώρα έχει το λόγο ο κύριος Ιλβα Περέιρα. Πρόεδρε, καταρχήν θα ήθελα να χαιρετήσω την ε, σύναψη της συμφωνίας με το Βιετνάμ που είναι σημαντικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική Ασία. Είναι μια συμφωνία νέας γενεάς, άρα πρότυπο για τις μελλοντικές συμφωνίες με τις χώρες ΑΣΕΑΝ. Αλλά ε, δεν είναι αυτός σκοπός η εμπορική συμφωνία αποτελεί μία στρατηγική θέση για να προωθήσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες και ιδιαίτερα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό και ανησυχούμε σε σχέση με την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ, ιδιαίτερα ως προς την ε, ελευθερία του εκφράζεστε. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε μία προσέγγιση ερεσιμότητας ως προς τις εμπορικές συμφωνίες. Θα ήθελα να ρωτήσω την Επίτροπο τι πρόοδος έχει επιτελεστεί στο Βιετνάμ ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα από την απαρχή των διαπραγματεύσεων και τι διδάγματα έχουμε να εξαγάγουμε από αυτή τη διαδικασία. Η συμφωνία με το Βιετνάμ πραγματικά τηρεί την αρχή της αιρεσιμότητας σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα σε μια εμπορική ατζέντα. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Επίτροπε. Θα ήθελα να πω ότι ως μόνιμος εισήγητη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου για την Εμπορική Συμφωνία με το Βιετνάμ δεν υποστηρίξα την κατάθεση της ε, προφορικής αυτής ερώτησης και τη συζήτηση αυτή στην Ολομέλεια. Παρ' όλα αυτά ήμουν ε, σε μειωτική θέση, μειοψηφική θέση στην Επιτροπή και το σέβομαι αυτό. Στις ε, διαπραγματεύσεις λοιπόν για την εμπορική αυτή συμφωνία δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα και πιστεύω ότι οι δεσμεύσει είναι επαρκής και ότι το Βιετνάμ θα εκπληρώσει τις δεσμεύσεις αυτές. Είναι δικό μας καθήκον άλλωστε να, να δούμε ότι εκτελούνται και ότι εφαρμόζονται αυτές οι δεσμεύσεις. Και τώρα είμαστε σε φάση οριστικοποίησης και ολοκλήρωσης αυτής της συμφωνίας και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γι' αυτό. Την άλλη εβδομάδα θα υπογραφεί η συμφωνία και θα ήθελα να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα φίλων του Βιετνάμ εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου εκπροσωπούνται όλες οι πολιτικές ομάδες. Και πιστεύω αυτό είναι μοναδικό και θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, η κυρία Γκίλ, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτροπή. Καλώς ορίζω αυτή την ε, Σύμφωνη Ελευθέρου Εμπορίου. Έχει πολλές δυνατότητες και ευκαιρίες ε, για την ανάπτυξη και για τις θέσεις εργασίες, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του τύπου, αλλά και για το Βιετνάμ. Αλλά αυτό το δυναμικό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον υπάρχουν τα σωστά μέτρα για να μεγιστοποιηθούν ε, τα θετικά, οι θετικέ συνέπειες και να μειωθεί η πιθανότητα των αρνητικών αντικτύπων είτε πρόκειται για τις διώξεις και τις ε, φυλακίσεις των αγροτών και όσων αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, η κατάσταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι θλιβερή στο Βιετνάμ. Γιατί λοιπόν δεν κάνει εξάντα αξιολογήση των ανθρώπινων δικαιωμάτων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι επίσης σαφές ότι τα συνήθιοι μέσα και εργαλεία δεν αρκούν στην προκειμένη περίπτωση γιατί έχουν και περιορισμούς οι οποίοι είναι ευρέως γνωστοί. Αλλά πώς μπορούμε τυφλά να εφαρμόσουμε μία τέτοια, τέτοια μέσα ελλειπή σε μία τόσο ευρεία συμφωνία ελευθέρου εμπορίου. Κάποιοι λένε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ένας μηχανισμός επικοινωνίας μεταξύ της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και του Κοινοβουλίου για την εφαρμογή των της συνεργασίας και της ανάπτυξης δυναμικού για να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Δεν προσπαθούμε να υπονομεύσουμε την Συμφωνία Ελευθερού Εμπορίου ή να δακτυλοδείξουμε την κυβέρνηση του Βιετνάμ, αλλά να τονίσουμε ότι η πρόληψη είναι πιο φθηνή και πιο αποτελεσματική από την, την, η θεραπεία και ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποια βασικά στοιχεία με τους στρατηγικούς μας εταίρους στην Ανατολική Ασία, ιδιαίτερα δεδομένη της κατάστασης. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Να περάσουμε στην διαδικασία Catch Έχουμε 7 άτομα που έχουν ζητήσει τον λόγο. Θα τους δώσω το λόγο, αλλά να τηρήσετε το ένα λεπτό. Ο κύριος Μπόκοβιτς καταρχάς έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν μια διαδικασία. Και η βάση λοιπόν για αυτό για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι να μην πεινάει ο κόσμος, να μην υποφέρει, να έχει μια παιδεία και εκπαίδευση και σε τελική ανάλυση αυτοί να απαιτήσουν και να προασπιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Η κατάσταση λοιπόν αυτή θα βελτιωθεί και είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι μετά τη συμφωνία αυτή ο κόσμος θα διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Όσοι πιστεύουν ότι σε ένα πολιτικό σύστημα όπου επικρατεί τέτοια φτώχεια, τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα σε υψηλό επίπεδο, θα πρέπει πολύ απλά να κάτσουν και να σκεφτούν. Τι γίνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ε, Λιβύη, στο Ιράκ και στη Συρία. Και σήμερα λοιπόν θα πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσον τηρούν τα ανθρώπινα δικαιώματα εκεί. Όχι βέβαια. Ακόμα και η ίδια η ανθρώπινη ζωή απειλείται. Τα ανθρώπινα δικαιώματα λοιπόν αποτελούν μια διαδικασία εν εξελίξη. Ο κ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Βρισκόμαστε σε ουσιαστικέ διαπραγματεύσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Βιετνάμ επέτυχαν μια συμφωνία για τι ελεύθερε εμπορικέ ανταλλαγέ και έτσι θα υπάρχουν ανταλλαγέ με μια πολύ δυναμική οικονομία τη Ασία. Μια συμφωνία η οποία θα είναι χρήσιμη και για τι δύο οικονομίε. Βεβαίω ε, είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι όσον αφορά την παραβίαση των δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. Έχουμε 24 ανεξάρτητε οργανώσει ε, και το μεγαλύτερο μέρο εταίρους της κοινωνίας των πολιτών επεξεργάστηκαν μια έκθεση που αφορά στην παραβίαση των δικαιωμάτων κατά το 2014. Εκεί λοιπόν περιλαμβάνονται παραβιάσεις για λόγους ε, θρησκευτική πίστης. Η συμφωνία ε, μπορεί να ανασταλεί σε περίπτωση ομής παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Κομισιόν θα πρέπει να επαγρυπνά σε μια ε, χώρα ε, όπως αυτή έτσι ώστε να επιτευχθεί μια βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για ένα λεπτό, ο κύριος Μαριάς. Με τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών που υπογράφτηκε τον Αύγουστο του 2015 ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Βιετνάμ εξαλείφονται οι τελωνιακοί δασμοί στο εμπόριο προϊόντων, υπηρεσιών και επενδύσεων και προβλέπεται αύξηση του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω του 2% στα πλαίσια των μεταξύ του διαπραγματεύσεων ευρωπαϊκή ένωση και βιετνάμ υποτίθεται ότι έχουν δρομολογήσει ένα διαρθρωμένο διάλογο που αφορά στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που πρέπει να είναι και η βάση κάθε εμπορικής συμφωνίας σύμφωνα με τη συνθήκη της ευρωπαϊκής ένωσης. ωστόσο η συμφωνία αυτή δεν δίνει δεκάρα για τι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που λαμβάνουν χώρα σήμερα στο βιετνάμ και κάνει όπως και οι άλλες εμπορικές συμφωνίες όπως είναι η ttip και η tisa το μόνο που τις ενδιαφέρει είναι να αποσκοπούν στην κερδοσκοπία των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων σε βάρος των μικρομεσαίων και έτσι οδηγούν στη μείωση της απασχόλησης στις χώρες που εφαρμόζονται. γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να έχουμε προώθηση συμφωνιών οι οποίες να μην πλήττουν την απασχόληση και τους εργαζόμενους και να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο κύριος Τσίτς, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ε, κύριε κυρία Πρόεδρε, με εκπλήσουν τα επιχειρήματα ορισμένων συναδέλφων. Λένε ότι δεν θα πρέπει να υπογραφεί αυτή η συμφωνία διότι δεν τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ξέρουμε ότι γενικά δεν ε, την χάνουν σεβασμού τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά δεν μπορούμε εμείς να επιβάλλουμε τη δική μας δημοκρατία, δεν μπορούμε να εξαγάγουμε τη δική μας δημοκρατία σε άλλες χώρες. Δεν είναι σωστή η λογική αυτή. Κυρία Επίτροπε, θεωρώ ότι ε, εμείς θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια στο Βιετνάμ το Βιετνάμ είναι μία από τις πιο φτωχές χώρες του κόσμου, γι' αυτό τάσουμε υπέρ της συμφωνίας, γνωρίζοντας ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Βιετνάμ ε, είναι ένα θέμα που παραμένει ανοιχτό. Αλλά θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή τη συμφωνία λόγω φτώχειας. Ο κύριος Σόγκορ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην ε, τήρηση και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναμφίβολα και αυτό θα πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη όταν συνεργαζόμαστε με τρεις ε, χώρες. Δεν θα πρέπει όμως να είμαστε ε, ιδεαλιστές με τη στενή έννοια και να λέμε ότι δεν θα δεχτούμε τη συνεργασία με χώρες που δεν έχουν μια εύρωστη πολιτική τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Φυσικά δεν είναι μια ε, χώρα προς μίμηση το Βιετνάμ, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε τη συνεργασία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολλές φορές είναι επιφυλακτική να καταπολεμήσει, να καταδικάσει πρακτικές σε τρίτες χώρες. Αυτό δεν ενισχύει την αξιοπιστία μας. Ο κύριος Φρουνζουλίκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Συμφωνώ ως προς την ανάγκη της στήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένα θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει την Επιτροπή κατά τις διαπραγματεύσεις με το Βιετνάμ για τη σύναψη συμφωνίας, ιδιαίτερα σε σχέση με την ελευθερία του εκφράζεσθε και του συνεταιρίζεσθε της, ε, το δικαίωμα στην ανεξιρθρησκεία, το δικαίωμα στην αντίρρηση γενικότερα. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη τα δεδομένα μελών της κοινωνίας των πολιτών και κοιό. Πιστεύω ότι οι συμφωνίες ε, ελευθέρου εμπορίου δείχνουν ότι έχουν και περιορισμούς, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την φιλελευθερωποίηση και την βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής που θα προωθήσει. Sorry, for one minute. Ναι, για ένα λεπτό ο κύριος Μικολασίτς έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπέ. Η συμφωνία αυτή με το Βιετνάμ, η οποία σχετίζεται και με την συνεργασία, με τη Συμφωνία Εταιρική Σχέση και Συνεργασία μπορεί να, να αποτελέσει υπόδειγμα για το πώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ζητήσει από τους νέου εμπορικού εταίρου εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και πιστεύω ότι είναι πραγματικά μεγάλη ανάγκη να κοιτάξουμε και τα άτομα με αναπηρία. Να δούμε τα άτομα τα οποία δεν μπορούν να συναθρίζονται γιατί δεν υπάρχουν ε, ανεξάρτητα Ινδικάτα, η Σαϊγκόνη, η οποία ήταν παράδειγμα στην χώρα και όπου υπήρχαν και συμβίωναν ελληνικά διάφορα θρησκευτικές κοινότητε, πλέον καταπιέζεται και έτσι λοιπόν θα πρέπει όλα αυτά να λεφτούν υπόψη στην εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας και να ασκηθεί πίεση προς τους εταίρους προκειμένου να τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ και έχετε τώρα το λόγο, λέει η πρόεδρο την κυρία Μάντουστρομ, για να απαντήσετε στη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Το εμπόριο μόνο του δεν μπορεί βέβαια να λύσει όλα τα προβλήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μπορεί όμως να συμβάλλει έτσι ώστε να ε, στηρίξουμε την ανάπτυξη και αυτό πρέπει να κάνουμε με τις συμφωνίες μας και κυρίως με αυτήν που συζητάμε σήμερα με το Βιετνάμ. Κανείς ε, δεν αρνείται ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Βιετνάμ. Είπατε πολλά, μπορώ και εγώ να προσθέσω άλλο. Υπάρχουν, είναι σοβαρά. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε ε, καθώς συζητάμε με τις αρχές του Βιετνάμ. Υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις, αλλά από ό,τι φαίνεται θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε τα απαραίτητα εργαλεία, έχουμε τη νομική σχέση ανάμεσα στην Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου και την Συμφωνία Συνεργασίας Partnership Agreement. Θα κάνουμε αξιολόγηση, κυρίως όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε τον διάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα υπάρξει μια σχετική συνάντηση και πάλι μετά από κάποιες εβδομάδες θα συστήσουμε ε, συμβουλευτικές ομάδες με την κοινωνία των πολιτών για να ε, μιλήσουμε επί τόπου με ανθρώπους που γνωρίζουν την κατάσταση. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε όλα αυτά να τα δημοσιεύσουμε μέχρι τέλος της εβδομάδας για να εξηγήσουμε πώς ακριβώς ε, τα μέτρα που υπάρχουν της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και τα μέτρα της Συμφωνίας Ελεύθερων Εμπορικών Ανταλλαγών θα συμβάλλουν στο να υπάρχουν να υπάρχει ελευθερία στα, και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και εν πάση περιπτώσει όλα θα αξιολογηθούν από τη στιγμή που θα τεθούν σε ισχύ. Όλα θα είναι διαφανή, να μπορείτε να ε, παρακολουθείτε το διάλογο. Υπάρχουν ε, βέβαια σαφείς ε, προϋποθέσεις, προαπαιτούμενο όπως λέγονται στη συμφωνία, αλλά επιθυμούμε να υπάρξουν συγκεκριμένα φόρουμ διαλόγου για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να επιτύχουμε κάποια βελτίωση. Δεν έχουμε καμία σημασία συμφωνία με το Βιετνάμ για αυτά τα φόρουμ και δεν είμαι σίγουρη κατά πόσον όλα αυτά θα δώσουν περισσότερα δικαιώματα στους Βιετναμέζους. Τελικά αυτή η συμφωνία θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Μετά από λίγο θα δημοσιευτεί να μπορείτε κι εσείς να τη δείτε, να κάνετε τη δική σας αξιολόγηση και βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει η μετάφραση, όλα αυτά τα νομικά διαδικαστικά. Θα υπάρχει αρκετός χρόνος για να συζητήσουμε και βεβαίως η Κομισιόν είναι πρόθυμη να ξεκινήσουμε το διάλογο. Για άλλη μια φορά σας λέω ότι θα σας κρατήσουμε ενήμερους. Ε, είμαστε στη διάθεσή σας για τις απόψεις σας για να έχουμε διάλογο μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε.